Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίαση με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έκθεση ε, του συναδέλφου κυρίου Λουίς Μανουέλ Καπούλα Σάντος με θέμα άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς. Ο εισηγητής, ο συνάδελφος κύριος Καπούλα Σάντος έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ε, να σας καλησπερίσω, όπως να καλησπερίσω και τον κύριο Επίτροπο και να εκφράσω την ικανοποίησή μου. Διότι σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό, ίσως να μην μου χρειαστούν καν τα τέσσερα λεπτά που μου δώσατε, διότι Νομίζω ότι έχουμε πετύχει συνένεση. Γνωρίζουμε πως η Επιτροπή της Κομισιόν είναι μια πρόταση που θέλει να εγγυηθεί τη συνέχιση των άμεσων ενισχύσεων σε αυτό το μεταβατικό έτος ανάμεσα στην σημερινή ΚΑΠ και την μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πολιτου προγράμμα, πλαισίου. Η πρόταση αυτή καθορίζει για το έτος 2013 και για το οικονομικό έτος 2014 τις εθνικές ε, επιδοτήσεις, ενισχύσεις μάλλον και το σύνολο των ποσών για τις άμεσες αυτές ενισχύσεις που λαμβάνουν υπόψη και την ε, ένταξη των νέων χωρών και να εγγυηθούν ένα μηχανισμό όπως αυτό της διαφοροποίησης για να εγγυηθούμε σταθερότητα στα ποσά που χορηγούνται στους γεωργούς τελευταίο έτος 2013 η Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου μας έχει προβλέψει ορισμένες νέες διατάξεις για συγκεκριμένες καταστάσεις που επικρατούν κράτη-μέλη με βάση τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Αναφέρουν στον Ενέν Βασίλειο, τη Γερμανία και την Σουηδία. Για το 2013 προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα για τα νέα κράτη να χρησιμοποιήσουν ή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν εθνικά ποσά του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ και προβλέπεται και μια ανάλογη διάταξη για την Κύπρο, κάτι το οποίο αποφασίστηκε στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Ε, τα αποτελέσματα του διαλόγου εστάλησαν στην Επιτροπή Γεωργίας και εκεί επιτεύχθηκε μια ευρύτατη συνένεση. Να ευχαριστήσω τι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προθυμία του, τη διαθεσιμότητά του, την ιδανική προεδρία του Συμβουλίου και να ευχαριστήσω την γραμματεία της Κομάγρη της Επιτροπής Γεωργίας. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής Γεωργίας, της Νομικής Επιτροπής και οι σκιώδεις ε, ασχολήθηκαν σε βάθο με το θέμα προκειμένου να υπολογιστούν τις εγγυήσει ε, για τις πληρωμές σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, αυτή τη μεταβατική χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ, κάνω έκκληση ε, να υπερψηφιστεί το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια προκειμένου να μπορέσει να δημοσιευθεί η λόγω νομοθεσία και να μπορέσουν αυτοί, αυτές οι πληρωμές να γίνουν εγκαίρως στους γεωργούς την προσεχή χρονιά. Ευχαριστώ για την προσοχή. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Ντάτσιαν Τσόλος εξ ονόματος Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε. Merci, euh, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι που βλέπω ότι η νομοθετική διαδικασία για την έγκριση της πρότασης Κομισιόν αναφορικά με τις άμεσες ενισχύσεις το 2013 βρίσκεται τώρα στην τελική φάση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάπουλα Σάντος, τον εισηγητή, αλλά και τον πρόεδρο ε, της Επιτροπής Γεωργίας, κύριο Παύλο Ντεκάστρο, για τις προσπάθειές τους προκειμένου να προχωρήσει αυτός ο φάκελος τάχιστα μέσω της διαδικασίας και την ε, ε, βούληση να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, κάτι που θα μας βοηθήσει να λάβουμε άμεσα απόφαση. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τάχιστη έγκριση αυτού του κανονισμού για να διασφαλίσει την καλή χρησιμοποίηση αυτών των ποσών το 2013. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εκφράζω την ικανοποίησή μου που το συμβαστικό κείμενο βρίσκεται στη μέση διάταξη αυτή τη ολομελία και θα ψηφιστεί αύριο το πλαίσιο του τριμερού διαλόγου, του άτυπου τριμερού διαλόγου που διεξήχθη στι 24 Μαου ενεστώτο έτου. Μια συμφωνή πολιτική επιτεύχθη με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί τη προτάσεω τη Κομισιόν. Το συμβαστικό αυτό κείμενο περιέχει μια σειρά τροπολογιών που κρίνονται απαραίτητε ε, με κοινή συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και η Κομισιόν της Προσυπογράφηση. Γνωρίζω επίση πω ορισμένα στοιχεία αυτή τη πολιτική συμφωνία έγιναν με βάση την αρχή ότι το πεδίο εφαρμογή αυτού του μεταβατικού του περιορίζεται το 2013 και δεν προδικάζει αποφάσει που θα ληφθούν στο πλαίσιο τη μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και τι δημοσιονομικέ προοπτικέ που ελπίζω να εγκριθούν όσο νου. Ε, τώρα δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Τζοβάνι Λαβία, εξ ονόματο τη Επιτροπής Προπολογισμών, για ένα λεπτό. Ουκ εν το πολλό το εφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και από πλευρά μου και από πλευρά τη Επιτροπή προπολογισμών. να πω ότι συμφωνούμε και χαιρόμεθα που αυτή η διαδικασία κλείνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, ένα ζήτημα μόνο που αφορά στην Επιτροπή Προπλοισμών και είναι η σχέση που οι άμεσες ενισχύσεις του 2013 έχουν σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως γνωρίζετε, η γεωργική χρονιά ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου και οι άμεσες πληρωμές που θα πρέπει να χορηγηθούν το 2013 θα αφορούν στον προπολισμό του 2014. Αυτό το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο δυστυχώς δεν ε, κάνει γοργαβήματα και το συμπέρασμα της ε, Δανικής Προεδρίας ήταν ε, το να, μεταθέ, να μεταθέσει αυτή την εργασία στην Κυπριακή Προεδρία που θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Ελπίζουμε το ζήτημα αυτό να ολοκληρωθεί το συντομό των δυναστών διότι όχι θα επιτρέψει τις άμεσες πλωμές μέσα στο 2013 αλλά και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης το συντομότερο των Ευχαριστώ ανοίγει ο κύκλος των, των <clears throat> εξ των πολιτικών ομάδων και πρώτη έχει το λόγο η συνάδελφος κυρία Μαρία Νεντέλτσεβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαίσια εργασία του. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διατυπώνει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι που κάνει τις προτάσεις, τις πληρωμές τις κατανέμει η Κομισιόν και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις νέες χώρες μέλη και εύχομαι να έχει πιο φιλόδοξους στόχους. Χρειαζόμαστε μια πιο δίκαιη κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, εφιστώ την προσοχή στο ρόλο των χωρών μελών οι οποίες είναι αυτές που μπορούν να εντοπίσουν τις ανάγκες των γεωργών στις χώρες μέλη. Να συνεργαστούν λοιπόν, αυτό του ζητώ, πιο ενεργά. Ένα σημαντικό μέρος της ε, νομοθετικής διαδικασίας του ανήκει, παρόλο που σήμερα δεν είναι παρούσες εδώ το Συμβούλιο δηλαδή. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς καλούμαστε να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα όλων και οριζοντίως και καθέτος. Ελπίζω και οι υπόλοιπε εκθέσεις σχετικά με την ΚΑΠ να δώσουν τα τελικά χαρακτηριστικά σε όλη την προσπάθεια. Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Ήβαρη ε, Πάνταρ, εξ ονόματος των, της των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω τις ε, τροπολογίες των εισηγητών και ιδίως εκείνες που δίνουν ευκαιρία στις νέες χώρες μέλη να ε, δώσουν εθνικές ενισχύσεις το 2013 διότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις θα διευκολύνουν το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων γιατί χωρίς αυτές τις συμπροματικές ενισχύσεις οι γεωργοί θα λάβουν περίπου 20% λιγότερη υποστήριξη. Πρόκειται για ένα λογικό συμβιβασμό που αποτελεί μια χρήσιμη αφετηρία για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την περίοδο 2014 έως 20 και είναι θετικό το μήνυμα που δίνεται έτσι στους ε, γεωργούς των βαλτικών χωρών ότι είναι δυνατόν, δηλαδή να ξεβρεθούν θετικοί συμβιβασμοί. Σειρά έχει τώρα εξ ονόματος της ομάδος ALDE η συνάδελφος κυρία Μπρίτα Ράιμερς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κύριε και κύριοι. Από την ομάδα των φιλελευθέρων εμείς υποστηρίζουμε τις τροπολογίες. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι με τον συμβασμό στον οποίο καταλήξαμε και με την διατήρηση των εξωτερικών εξαιρετικών περιστάσεων επιτρέπεται να δοθούν ενισχύσεις στους γεωργούς. Είναι σημαντικό στο μεταβατικό αυτό έτος να έχουμε ξεκάθαρες θέσεις. Επίσης τονίζω τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε και εκφράζω την ευχή αυτή η επικοδομητική συνεργασία να συνεχιστεί και στο μέλλον, διότι μέχρι τώρα σκόνταψε σε πολλές φάσεις η κοινή αγροτική πολιτική. Ελπίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να συνεργαστούμε για να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα υπέρ των Γεωργών. Thank you, Mr. Reimers. On behalf of the Green, one minute and a half speech time for our colleague Anna Miranda. Obrigada, Obrigada. Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κάπουλα Σάντος, ο οποίος ε, πάντα ε, ήταν υπέρμαχος της Γεωργίας και ελπίζουμε να συνεχίσει και στο μέλλον έχοντας υπόψη την μετέθμιση της ΚΑΠ γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση των γεωργών που προσδοκούσαν αυτήν την συνέχιση των ε, άμεσων ενισχύσεων. Θα ήθελα να αναφερθώ στην χώρα μου, την Γαλλικία. Είναι μια αγροτική περιοχή επαντηλημένα μας έχει απασχολήσει. Ο προϋπολογισμός ε, και η χρηματοδότηση είχε παγώσει για τα θέματα της ε, αγροτικής ανάπτυξης λόγω ακριβώς ε, των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι άμεσες ενισχύσεις. Αυτός ο κανονισμός βασίζεται σε μια συνένεση που επιτεύχθηκε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε, μια στιγμή που ο γεωργικός τομέας ε, γνωρίζει σοβαρή κρίση διότι ε, απουσιάζει η δημόσια στήριξη του κλάδου. Αυτή η προσαρμογή σχετικά με την διαφοροποίηση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Να υπενθυμίσω την ελληπή πρικοδότηση που προβλέπεται για την μελλοντική μεταρρύθμιση η οποία θα μειώσει σημαντικά το ποσοστό της χρηματοδότησης ε, μέσω του εθνικού προπολογισμού. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και αυτό υπόψη μας. Ευχαριστώ. ECR, ε, το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κ. Γιάννος Βοησεκόφσκι. Για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα τον εισηγητή κύριο Κάπουλα Σάντος για την εργασία του, για το γεγονός ότι μέχρι το 2020 οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, κάτι που χρειάζεται τόσο πολύ. Ελπίζω το έτος 2013 να είναι το τελευταίο έτος όπου στις άμεσες ενισχύσεις θα σημειωθούν τόσο μεγάλες διαφορές προ περίπου προσθέθηκαν νέες χώρες μέλη στην Ένωση και οι αγρότες κατάλαβαν τότε ότι θα καλούνταν να εργαστούν και να αποδώσουν μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με άνισους όρους ανταγωνισμού. Τώρα λίγη αυτή η περίοδος, ενώ βέβαια για τη Βουλγαρία και η Ρουμανία θα συνεχιστεί ακόμη. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Σάντος. Μετά από το 2014 ελπίζω ότι δεν θα υπάρχουν πλέον διακρίσεις σε ό,τι αφορά την καταβολή των άμεσων ισχύσεων. Ε, της ΓΚΟΕ είναι ο συνάδελφος κύριος για λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύουμε ότι το 2013 θα ληφθεί ως ε, έτος αναφοράς βέβαια για τον πολιετή σχεδιασμό για τις καταβολές αυτές που είναι πολύ σημαντικές για να εξισώνονται οι όροι ανταγωνισμού. Η δική μου πολιτική ομάδα και οι γεωργοί της Λετωνίας θεωρούν ότι είναι απαραίτητες οι άμεσες ενισχύσεις για να εξισώνονται, να εξορροπούνται οι όροι ανταγωνισμού στην αγορά, αλλά και για να αποδίδεται κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι ορθό το περιεχόμενο της εκθέσεως Κάπουλα Σάντους. Και σέβομαι βεβαίω και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να ανέρχονται στο 80% του αγροτικού προϋπολογισμού. Τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μόνο για δικαιοσύνη γιατί οι βαλτικές χώρες λαμβάνουν πολύ λιγότερα αναλογικά από τις ε, άμεσες ενισχύσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα λετονοί γεωργοί να εγκαταλείπουν την ύπεθρο της χώρας και να αγοράζουν τα κτήματα άλλοι, αλλοδαποί και καταστρέφονται έτσι τα κτήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγή για όλη τη δουλειά του και για την πρόοδο που έχει επιτύχει σε σχέση με το θέμα ε, των αμέσων πληρωμών για το 2013. Βεβαίως είναι σημαντικό να προβλέψουμε τις πληρωμές αυτές για το 2013, αλλά πρέπει να προβλέψουμε και για την ανάπτυξη την αγροτική και αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ σημαντικό. Ακόμη Σπουδαίο είναι για μας ότι υπάρχουν δεσμεύσεις πληρωμών για λιγότερο ε, ευνοούμενες περιοχές και διάφορα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης. Ακόμη, σημαντικό είναι η μεταβατική περίοδος για αυτές τις πληρωμές να είναι ομαλή και περιορισμένη όσον αφορά την επίδραση στο εισόδημα των γεωργών, ιδιαίτερα λόγω της ασάφειας της παγκόσμιας αγορά, αγορές. Ελπίζω ε, να προχωρήσουμε λοιπόν επικοδομητικά. Η κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013 πρέπει επίσης να αναγνωρίσει την ανάγκη άμεσων πληρωμών και να υποστηρίξει αυτούς που είναι ενεργοί γεωργοί και παράγουν ασφάλεια τροφίμων στην Ευρώπη. Ε, οι πληρωμές του πυλώνα 1 πρέπει να αναγνωρίσουν το χρόνο που καταναλώνουν οι γεωργοί για να παράγουν τρόφιμα και ο πυλώνας 2 παράγει αν θέλετε καλύτερες πληρωμές για την ένταξη μέσα στο περιβάλλον. Ακόμα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί στο να έχουμε μια λογική ρύθμιση μέσα στο πολιετές και να διορθώσουμε ανισορροπίες στις ε, κατανομές, στην γεωργική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει ε, πολύ κακή ε, κατανομή και πρέπει να λυθούν οι ανισορροπίες. Συνάδελφοι, για τήρηση του χρόνου ομιλίας, ε, τώρα ανοίγουν, ακολουθούν οι λοιποί εγγεγραμμένοι ομιλητές και δίνω μέσα το λόγο στον συνάδελφο κύριο Νικουλέσκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση για άμεση ενισχύσει το 2013 προς τους Γεωργούς αποτελεί το νομικό πλαίσιο. Η προτάσεις και της ε, Κομισιόν και, του εισηγητού είναι δίκαιες και ισορροπημένες και για τη Βουλγαρία και για τη Ρουμανία. Διότι η, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια η σταδιακή εφαρμογή των ε, ενισχύσεων αυτών και η Ρουμανία δεν υπάρχει ακόμα ε, οροφή. Κάτι το οποίο βέβαια είναι δίκαιο. Έτσι το Κοινοβούλιο πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα προς την κατεύθυνση της, ε, του σχεδιασμού της επόμενης κοινή αγροτικής πολιτικής. Σύντομα βέβαια θα, συζητούμε, θα συζητήσουμε και τις επόμενες εκθέσεις στην ε, Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων και θα τα, θα τα συζητήσουμε βέβαια το κάθε πράγμα στον καιρό του. Στο μέλλον θα πρέπει να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να φτιάξουμε ένα δίκαιο σύστημα που να επιτρέψει στη Ρουμανία και Βουλγαρία να εισαγάγουν στα, στα, σταδιακά. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Ούλρικε Ρόντουστ. Äh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κύριε και κύριοι, βρισκόμαστε μέσα στην διαδικασία της διαμόρφωσης αγροτικής πολιτικής. Το ΔΕ Κοινοβούλιο αύριο θα ψηφίσει το πρώτο σχέδιο κανονισμού για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων για το μεταβατικό έτος 2013. Και καλώς. Και μάλιστα αυτό είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή Λουίς Κάπουλα Σάντος για την ορθή, ξεκάθαρη και ταχεία εργασία του. Θα αρχίσουν να ισχύουν αυτά από το 2014 για να μην υπάρξουν προβλήματα στη μεταβατική περίοδο ήταν απαραίτητο να γίνει ταχεία συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η συνέχεια των χρηματοδοτήσεων είναι κρίσιμη για τις χώρες μέλη και γι' αυτό είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν σωστά οι ρυθμίσεις για το μεταβατικό έτος 2013. Ορισμένες από τις ρυθμίσεις όμω περιλαμβάνονται στα κείμενα ισχύουν μόνο μέχρι το 2012. Χαίρομαι πάντω που έχει εξευρεθεί λύση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και κυρίω για να γίνουν οι μεταφορέ από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Συνάδελφος Άλιν Σμιθ για 1,5 λεπτό. Thank you, President. Uh, I'll be uh, no exception in uh, congratulating. Και εγώ θα συγχαρώ βεβαίω ε, τον δυναμικό μα, εισηγητή Λουίς για την καλή δουλειά που υποβάλλει σήμερα και χαίρομαι που τα κατάφερε, αλλά είναι καλή δουλειά που έχει κάνει και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν για να εξασφαλίσουν κάποια σαφήνεια που είναι σημαντική όπως για τα ε, προγράμματα ανάπτυξης της ε, υπαίθρου για τις ε, περιοχές οικολογικής στόχευσης και ούτω καθεξής. Ας μην λησμονούμε ότι το θέμα υπό ορισμένε περιστάσει και περιστάσεις και ορισμένου κύκλου είναι επίμαχο. Υπάρχουν χώρε μέλη οι οποίε επιθυμούν να μειώσουν, να περικόψουν τι άμεσε ενισχύσει. Ενώ τουλάχιστον από τη σκοτσέζικη πλευρά είναι απαραίτητε για την, ε, για την ε, αγροτική οικονομία. Χαίρεται λοιπόν η σκοτική κυβέρνηση που συνεχίζουμε έτσι. Και είναι ατυχές ότι η χώρα μέλος στην οποία βρισκόμαστε έχει παίξει λιγότερο επικοδομητικό ρόλο. Πάντως κύριε Επίτροπε και στα Βρετανικά νησιά έχετε κάποιους συμμάχους οι οποίοι θα αγωνιστούν μαζί σας για τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Στη συνάδελφο κυρία Γκέρλινγκ για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καλωσορίζω την υποστήριξη των μελών της Επιτροπής Γεωργίας και ελπίζω και στην Ολομέλεια για αυτή την εθελοντική διακύμανση. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο τέλος της ουράς όσον αφορά την κατανομή της ΚΑΠ. Παρά αυτή την κακή διευθέτηση, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε πολύ σημαντικά σχέδια για το περιβάλλον της γεωργίας. Δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή με τους γεωργούς και δεν είναι και ο άμεσος τρόπος συνέχισης αν θέλετε, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε μέσω των αμέσων ενισχύσεων τη σταθερότητα για αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Καπούλα Σάντος για την ρεαλιστική προσέγγιση του και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Πατρίκ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Καπούλα Σάντος για το έργο του. Η μεταβατική πρόταση που μας έχει υποβληθεί είναι λογική, την υποστηρίζουμε. Έστω και αν αντιτίθεμε στο, από, συνδεδεμένε πληρωμές και την ενίσχυση βάση της εδαφικής τραυματικής έκτασης. Καλύτερα να ενισχύουμε την εργασία και όχι τη βιομηχανική γεωργία. Υποφελούμε από την ευκαιρία για να σας πω ότι μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ πρέπει να συζητήσουμε και το προσδιορισμό βασικών τιμών ε, με διακύμανση των ενισχύσεων ανάλογα με τις γεωγραφικές, τα γεωγραφικά δεδομένα, την απασχόληση κτλ. Θα χρειαστεί επίσης να υποστηρίξουμε τον ε, προϋπολογισμό της ΚΑΠ για τα εισοδήματα των γεωργών και για ε, την κοινωνική δικαιοσύνη. Ε, τώρα στο βήμα την συνάδελφο κυρία Νικόλ Σινκλέρ για ένα λεπτό. Thank you, Mr. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί από τους πολίτες μας θεωρούν ότι βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις. Οι άμεσες ενισχύσεις είναι τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού που είναι το 40% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά χρήματα. Η συντηρητική κυβέρνηση ε, δεν χρησιμοποιεί ορισμένες ε, από αυτά τα κονδύλια για την υποστήριξη των γεωργών. Ουσιαστικά δημιουργούν ανισορροπίες μέσω εθελοντικής μείωσης της, των αμέσων ενισχύσεων γρηγορότερα από άλλα κράτη ε, μέλη. Γι' αυτό θα είμαι ε, κατά των τροπολογιών 1, 12 και 13. Οι γεωργοί της Ηνωμένας ε, Βρετανίας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω διακριτικής μεταχείρισης προς το Ηνωμένο Βασίλειο χρειαζόμαστε σωστή κατανομή των κονδυλίων από τον πυλώνα 2. Και τελευταίος ομιλητής, ο συνάδελφος κύριος ε, Ταμπάτζη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή Κάπουλα Σάντος για την θαυμάσια δουλειά που έκανε και που επιτρέπει να συνεχιστούν οι άμεσες ενισχύσεις χωρίς να μειωθούν το 2013 στις νέες χώρες μέλη. Φτάσαμε επιτέλους σε ένα επίπεδο όπου εξισώνονται οι πληρωμές στις παλαιές και στις νέες χώρες. Βέβαια, χαίρομαι που ο κύριος Κάπουλα Σάντος κατενόησε το πρόβλημα που θα προέκυπτε από το 2014 και μετά όταν θα λάβουμε νέα βάση για τις ενισχύσεις. Διότι ισχύουν αυτά που προβλέπουν οι παράγραφοι ε, Β και Γ του άρθρου 61 για εθνικές ενισχύσεις. Ο εισηγητής δικαίως εντόπισε το πρόβλημα ότι δηλαδή δεν επιτρέπεται να υποστούν δυσμενή διάκριση οι νέες χώρες μέλη. Και παρακαλώ κύριε Επιτρόπε να... Τώρα ανοίγει η διαδικασία Catch the Eye και καλώ στο βήμα τον ε, συνάδελφο κύριο George Lyon. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με κάποια ανησυχία και στο Λονδίνο και στο Holbridge όταν δημοσιεύτηκαν οι νομοθετικές προτάσεις του Επιτρόπου μας ανησύχησαν διότι δεν υπήρχε η θελοντική διακύμανση. Και στην Αγγλία και στη Σκωτία χωρίς τη δυνατότητα να αλλάξουμε την κατεύθυνση των ε, κονδυλίων προς την αγροτική ανάπτυξη θα είχαμε τεράστιες μαύρες τρύπες ε, για το έτος 2013 σε αυτά τα προγράμματα. Ευτυχώς η πίεση από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τις σκοτικές αρχές και με τη βοήθεια των συναδέλφων στο Ευρωκοινοβούλιο Τζακ Νίκολσον, Σάντο κτλ. Μπορέσαμε να τα ξαναβάλουμε στο πακέτο και θέλουμε κάποιε διαβεβαιώσει ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Σκοτίο θα μπορούν η κυβέρνηση να αποφασίσει εάν ε, θέλουν να μετακινήσουν τα κονδύλια χωρίς να έχουμε αυτές τις μεγάλες μαύρες τρύπες στην χρηματοδότηση το 2013. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη βοήθεια που έλαβα και ελπίζω και τα επόμενα δύο νομοθετικά πακέτα να περάσουν εύκολα, αν και αμφιβάλλω συνάδελφο Σόνικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το περιεχόμενο της εφιούς αυτής εκθέσεως και με την ευκαιρία θα, πω το εξή. Σε μια μελλοντική Ευρώπη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο ταχύτητες διότι θα υπάρξουν δύο ταχύτητες εάν δεν εξισώσουμε τις ενισχύσεις, τις καταβολές για όλες τις χώρες μέλη. Χώρες όπως η Σλοβακία αλλά και άλλες συνέβαλαν και αυτές στην προσπάθεια διάσωσης των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην δυσμονούμε λοιπόν ότι η αλληλεγγύη πηγαίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις. colleagues, I welcome this proposal, αυτή την πρόταση που είναι διοικητική αλλά δίνει στους γεωργούς κάποια βεβαιότητα για το επόμενο οικονομικό έτος. Έχω κάποια σχόλια να κάνω σε σχέση με τι άμεσε ενισχύσει προ του γεωργούς μετά το 2014. Είχα συναντήσει με διάφορου πολίτε τη περιφέρειας μας όσον πρέπει να εξετάσουμε τις μεταβολές στην έκθεση Κάπλος Σάντος. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη συνδεδεμένη βοήθεια. Ε, το πρασίνισμα επίσης είναι πολύ σημαντικό για να αλλάξουμε τις καλλιέργειες, αλλά δεν είναι πρακτικά αυτά που προτείνονται για τους μικρομεσαίους γεωργούς. Όσον αφορά τα οικολογικά θέματα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα ποσοστά να είναι εφαρμόσιμα και λεπτομερή και όσον αφορά τέλος τη σύγκληση, ε, χαίρομαι για την ε, σύζεξη που έκανε ο κύριος Κάπλο Σάντος ε, με τις προτάσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Συνάδελφος κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ουαλία η περιφέρεια μου εξαρτάται από τη Γεωργία. Ε, ε, συμβάλλει πολύ στην οικονομία της Ουαλίας. Ε, στις μειονεκτικές περιοχές όμως οι γεωργοί εξαρτώνται πάρα πολύ από τις άμεσες ανισχύσεις. Χωρίς αυτές τις ανισχύσεις πολλές οικογένειες θα εγκαταλείψουν τη γεωργία. Γι' αυτό χαίρομαι που συνεχίζονται αυτές οι άμεσες ανισχύσεις ιστορικά για το επόμενο έτος, ώστε να έχουμε την επόμενη ΚΑΠ. Θα ήθελα οι μεταβατικές ρυθμίσεις όμως να είναι ευέλικτες και να επιτρέπεται και η περιφερειακή ερμηνεία καθώς προσαρμόζονται οι γεωργοί μας. Και θα ήθελα ο Επίτροπος να έρθει στο Royal Well Show για να συναντήσει τους γεωργούς μας απευθείας. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Σιεκέρσκι. Ευχαριστώ. Το 2013 θα είναι έτος μεταβατικό διότι τότε λύγει το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013. Ήδη όμως τα βλέμματα είναι στραμμένα στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Χαίρομαι πάντως για την υποστήριξη προς τις εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν άνω των 5.000 ευρώ γιατί στις χώρες μας δίνονται λιγότερες άμεσες ενισχύσεις. Θα ήταν σωστό να βρεθούν και άλλες μεταβατικές λύσεις που να περιληφθούν στον κανονισμό, ώστε να ισχύσουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των νέων χωρών μελών και των παλαιών. Δεν θα έχουμε πλέον τομεακή στήριξη από το 2013 και μετά. ο τρόπος με τον οποίο θα καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις από το 2013 και μετά σημαίνει ότι ακόμη θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δηλώνω ιδιαίτερα ικανοποιημένος που εξευρέθη συμβιβασμός και ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Σάντος που πρότεινε θετικές λύσεις. Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε λοιπόν την διαφοροποίηση, θα μπορέσουμε μάλιστα να υποστηρίξουμε τους γεωργούς και στις παλαιές χώρες Η συζήτηση δείχνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις για όλους μας είναι σημαντικό εργαλείο στήριξης της αγροτικής οικονομίας. Διότι στο κάτω της γραφής οι αγρότες παράγουν για το κοινωνικό σύνολο, για το κοινό καλό και έχουν ανάγκη από σωστές τιμές και των μικρών χωρών οι γεωργοί έχουν ανάγκη από καλές τιμές όπως έχουν οι των μεγάλων χωρών η Γερμανία, η Γαλλία ας πούμε διότι στο κάτω της γραφής και αυτοί πρέπει να πληρώσουν τα λοιπάσματα για παράδειγμα στις ίδιες τιμές έτσι λοιπόν οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αφορούν μόνο τις παλαιές ή μόνο τις νέες χώρες μέλη υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των παλαιών χωρών μελών. Οι αγρότες στην Γαλλία έχουν διαφορετικές πληρωμές από άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή και του λέω όπως είπε και κάποιος άλλος ότι καλά τα πήγες και α χαρεί σήμερα γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει στι επόμενες εβδομάδες και μήνες. Πάντως καλύπτεται η κατάσταση διότι αλλιώς θα ήταν καταστροφή και ευτυχώ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε το δικαίωμά του να εξασφαλίσει ότι θα μπορούσαμε να καλύψουμε τα κενά που είχαν υπάρξει στο παρελθόν. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ η διαφοροποίηση, αλλά ήταν απαραίτητο να γίνει για να υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα και οι δεσμεύσεις, ιδίως στο Ενωμένο Βασίλειο. Και δεν είμαστε διόλου ικανοποιημένοι με τον δεύτερο πυλώνα που μας περιορίζει στο να προχωρήσουμε στην υλοποίηση καλών έργων. Ελπίζω η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μέσα σε αυτά δηλαδή, το, το Ηνωμένο Βασίλειο θα χαίρει και αυτό δίκαιο μεριδίου.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 mais aussi κάτι το οποίο μας επέτρεψε να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ρύθμιση για το 2013 για τις ε, άμεσες ενισχύσεις και για την ε, περαιτέρω ενίσχυση της γεωργικής ανάπτυξης, της αγροτικής ανάπτυξης. Ορισμένοι αναφερθήκατε σε κάποια σε εργασίε που προχωρούν και που αφορούν την μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική για την προσοχή ε, περίοδο δημοσιονομική. Παρακολουθώ τι ε, εργασίε ε, τη Επιτροπή Γεωργίας με βάση τις εκθέσεις των εισηγητών και ελπίζω σύντομα να ξεκινήσουμε και τις ουσιαστικές συζητήσεις με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για ε, να καταλήξουμε σε μια μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική που θα είναι πιο δίκαιη ε, βασιζόμενη σε μια σημαντική ε, στήριξη και χρηματοδότηση μέσω του προπολογισμού. Δευτερολογία του συναδέλφου του, του εισηγητού του κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα ευγενικά τους λόγια. Να ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο. Ε, πω ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να δουλεύουμε και να επικεντρωνόμεθα σε ένα ζήτημα που απασχολεί όλους μας. Όταν λοιπόν εστιάζουμε σε ένα κοινό στόχο μπορούμε ακόμα και τα βουνά να μετακινήσουμε αγωνιστήκαμε για κάποιο περίοδο, αλλά μπορέσαμε να επιλύσουμε προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το επικοσμητικό πνεύμα τόσο στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας αλλά και στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ελπίζω πως αυτό το θετικό κλίμα να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τις μελλοντικές μας εργασίες. Να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα σίγουρα θα πετύχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα στον τομέα της γεωργίας. Συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι. Το επόμενο, το επόμενο σημείο στην ε, ημερήσια διάταξη